Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε. Συνεδρία της Επιτροπής. Για να προκάνουμε. Να καλύψουμε τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, όπως καλωσόρισα και τους συντονιστές προηγουμένως, ακριβώς πριν που συνεδρίασαν, και θα ήθελα να καλωσορίσω όλα τα μέλη μας, τους αξιότιμους και αξιότιμες συναδέλφους μέλη της Επιτροπής μας. Επανακάμπτουμε μετά τη θερινή παρένθεση του Αυγούστου, διακοπές που ελπίζω να ξεκουραστήκατε να ανακτήσετε δυνάμεις όλοι σας και ελπίζω να φορτώσετε και πάλι τις μπαταρίες σας για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα. Το έργο μας με αφοσίωση ε, εντατικά και με πνεύμα καλής συνεργασίας και με θετική στάση και συμπεριφορά. Έχουμε πολλή δουλειά από σήμερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και βαριά η μερίσια διάταξη σήμερα. Αυτή τη βδομάδα συνεδριάζουν οι πολιτικές ομάδες κανονικά. Αλλά χρειάστηκε να συγκληθεί και συνεδρίαση της δικής μας πολιτικής ομάδας, γιατί, επιτροπής, συγγνώμη, ε, γιατί έχουμε ιδιαίτερα θέματα να εγκρίνουμε. Λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να εγκρίνουμε τη ημερήσια διάταξη. Αν δεν διαφωνείτε, θεωρείται εγκεκριμένη. Σημείο δεύτερο, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Θα ήθελα να σας πω ότι οι συντονιστές πρότειναν να οριστεί ο κύριος Δίας εισηγητή στο θέμα της απελευθέρωσης των διαβατηρίων με την Ταϊβάν, ε, η κυρία Ματιού, ε, εισηγήτρια για το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα πυροβόλα όπλα, εφαρμογή του άρθρου 10, και ο κύριος Μωράης, ε, εισηγητή για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ισλανδίας και Νορβηγία στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αμοιβαία δικαστική συνδρομή, σε ποινικά ζητήματα. Κλοντ, συγχαρητήρια. Χαιρόμαστε όλοι. Μ' αρέσει μέχρι τώρα η σταδιοδρομία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέει ο κύριο Μωράη. Και εμά. Χαιρόμαστε κι εμεί. Αν δεν διαφωνείτε, ορίζονται ε, οι τρει ε, συνάδελφοι εισηγητέ για τα θέματα που σα ανέφερα. Επίση, θα πρέπει να σα πω ότι η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθεσε υπόψη των οργάνων του Κοινοβουλίου την πρόταση του χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων για το έτος 2011 και ε, λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα αυτό τη ε, διαθεσιμότητα αιθουσών συνεδριάσεων και διευκολύσεων διερμηνίας για την Επιτροπή μας. Είναι πολλές συνεδριάσεις, πολύ εντατική οι ρυθμοί, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε και αίθουσες και προσθέτω, όσο γίνεται θα περιορίσουμε ε, τις συνεδριάσεις μας τη Δευτέρα και την Πέμπτη το απόγευμα συνήθως για να μπορέσουν να ταξιδεύουν τα μέλη της Επιτροπής και να φτάνουν. Θα προσπαθήσουμε στο βαθμό του δυνατού να συνεδριάζουμε αν χρειάζεται Πέμπτη, την Πέμπτη το πρωί για να μπορούμε να ταξιδεύουμε την Πέμπτη το απόγευμα. Ωραία. Σημείο τρίτο έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που βλέπετε στους φακέλους σας. Εάν δεν διαφωνεί κανείς, με τα πρακτικά. Ποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Κλάης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου ήθελα να αναφερθώ. Αν κατάλαβα καλά, ένα σημείο ε, στην ημερήσια ένταξη των συντονιστών ήταν το νέο σύστημα πόντων για την κατανομή των εκθέσεων. Το συζητήσατε αυτό στη συνεδρίαση των συντονιστών και παρακαλώ τι αποφασίσατε. Αλλάζει το σύστημα που ισχύει, θα μπορούσατε ίσως να μας ενημερώσετε σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι κύριε Κλάις, έχετε δίκιο. Μόλις ε, συνεφρίασαν οι συντονιστές και εγκρίθηκε αυτό το θέμα χωρίς αντίρρηση. Είχε συμφωνηθεί ε, προηγουμένως ε, κανονικά ισχύει το σύστημα DONT για τη διάθεση των εκθέσεων με βάση κάποιους πόντους. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό. Συνεχίζουμε όπως και στο παρελθόν με την ίδια μέθοδο για την ανάθεση των εκθέσεων για τις εκθέσεις συναπόφασης, τις διεθνείς συμφωνίες και άλλες εκθέσεις. Ακολουθούμε το συνήθες σύστημα. Εγκρίθηκε αυτό το σήμερα. Κύριε Κλάης, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω μια ερώτηση συγκεκριμένη για κάποιες εκθέσεις όπου δεν ενδιαφέρεται καμία πολιτική ομάδα. Γιατί ίσχυε ο εξή κανόν. Αν δεν ενδιαφέρεται καμία ομάδα και δεν είναι πρόθυμη να πληρώσει κανένα πόντο, οι μη εγγεγραμμένοι δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να λένε τη γνώμη τους. Δεν τους ρωτάει ποτέ κανείς αν ενδιαφέρονται να πάρουν τις εκθέσεις που δεν θέλει καμία πολιτική ομάδα. Και είναι ένα πρόβλημα και δεν μπορούν οι μη εγγεγραμμένοι να γίνονται εισηγητέ ποτέ. Στο μέλλον μπορείτε σας παρακαλώ να μας ρωτάτε και εμάς μήπως θέλουμε να πάρουμε καμία έκθεση. Είναι ένα θέμα που ήδη συζητήσαμε στην αρχή της θητείας, όταν έγινε η σύσταση των επιτροπών. Το συζητήσαμε ενδελεχώς και είπαμε ότι όταν δεν ζητηθούν εκθέσεις από τις ομάδες, τότε δεν έχουν πόντους. Και, εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση των μη εγγεγραμμένων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνένεση των συντονιστών, διότι ούτε η Προεδρία ούτε οι, επιτροπή, οι Επιτροπές στις κανονικές τους συνεδριάσεις μπορούν να το κάνουν. Μπουζούτιλ. Θα ήθελα επ' αυτού να πω κι εγώ κάτι. Εάν καμία πολιτική ομάδα δεν επιθυμεί μία έκθεση, τότε αποδίδεται στις ομάδες που δεν διαθέτουν πόντους. Αλλά σε ορισμένες περιστάσεις, εγώ συνάντησα μία ως συντονιστής του ΕΛΚ, όπου μονομερός οι ομάδες ε, δεν δέχτηκαν να αναλάβουν την έκθεση και την ανέθεσαν στους μη εγγεγραμμένους, έτσι ώστε και οι μη εγγεγραμμένοι να θεωρήσουν ότι συμμετέχουν στις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Το ΕΛΚ το έκανε μία φορά, δηλαδή απαρνήθηκε μία έκθεση, ελπίζω να γίνει και από τις άλλες ομάδες κάτι τέτοιο. Δηλαδή και άλλες ομάδες να σταθούν εξίσου γενναιόδορες. Σας ευχαριστούμε πολύ και όπως είπα και προηγουμένως, όταν δεν είναι επιθυμητές οι εκθέσεις, τότε δεν υπάρχει σύστημα πόντων. Το κανονικό μας σύστημα δηλαδή. Προσφεύγουμε σε αυτή τη ε, διαδικασία. Υπάρχει αυτή η, ε, η σύμβαση, δηλαδή να μην σπαταλώνται πόντοι. Αλλά είναι πολύ σκόπιμο αυτό που είπε ο κύριος Μπουζούτιλ. Άλλα σχόλια. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι νέο μέλος εδώ, αλλά μου φαίνεται περίεργο αυτό ότι δεν έχουμε Πόντου και εμείς εκλεγμένα μέλη του Κοινοβουλίου είμαστε. Πώς έχει ρυθμιστεί αυτό. Και κάτι άλλο που βρίσκω εξωφρενικό είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε καν παρόντες στη συνεδρίαση των συντονιστών. Για να σας πω το βρίσκω μέχρι και ηλίθιο αυτό το σύστημα. This point has been... Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί επί μακρόν και πολλές φορές δεν έχει νόημα να παράγουμε συζητήσεις, να επαναλαμβάνουμε συζητήσεις συζητήθηκε στην αρχή της θητείας ένα χρόνο πριν αλλά ο κύριος Άλβαρο ζήτησε το λόγο από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ. Εν κατακλείδη Σάιμον, δώσε μας μερικούς πόντους σας και θα τις ε, δώσουμε σε άλλους. Μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, γιατί εγώ έχω ένα φωτάκι κόκκινο που αναβασβήνει και δεν ξέρω κατά πόσο το σύστημα λειτουργεί. Are you asking, are you asking for... Δηλαδή θέλετε τεχνική βοήθεια, τι ζητάτε ακριβώς. Let me see, let me see, let me see. Let me see, just, just, just a second. I think, I think we all need to resort to electronic cards. Ναι, βγάλτε τις κάρτες σας για να κάνουμε έναν έλεγχο, να δούμε κατά πόσο λειτουργεί το σύστημα. Yep. Yes. Shall we go for a try vote? Ωραία. Κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Δοκιμαστική. Is it working? Ε, λειτουργεί. Εντάξει. Did it work? πράσινοι. Τρεις υπέρ πάνω από τον αριθμό, τον επιτρεπτό. Αυτό αφορά τους πρασίνους. Πώς και έτσι. Shall we... Θέλετε να ξαναδοκιμάσουμε. Αρχίζουμε πάλι τώρα δοκιμαστική. Βρεμόν. Apparently to our recording system. Σύμφωνα με το σύστημα καταγραφής έχουμε τρεις επιπλέον πράσινους. Και ένας επιπλέον μη εγγεγραμμένος. Αυτό πώς σας φαίνεται. <laughs> How about Please the mic. I mean, how many how many non have the right to vote in the? Πόσοι πράσινοι μπορούν να ναι. ψηφίσουν δύο. Και πόσοι μία εγγεγραμμένοι. Δύο. Εγώ είμαι ο τρίτος, αλλά είμαι ένα πρωτής. The, the problem is the system. Α, το πρόβλημα είναι το σύστημα. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα, τότε θα πρέπει να κάνουμε ειδική έκπτωση. Ε? Ε? Λοιπόν, σε περίπτωση αμφιβολίας θα σας μετρήσουμε ξεχωριστά. Σηκώνετε χέρια, εντάξει. Well, well, well, we have covered the preliminary points. Let's, let's go. Εάν έχουμε καλύψει τα βασικά, ας δούμε τα ουσιώδη. Η θέση του Κοινοβουλίου ως προς τον προϋπολογισμό του 2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το Συμβούλιο. Κυρία Ιντβέλτ αναλαμβάνει αυτό το σημείο, την ψηφοφορία δηλαδή. Okay, Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Θα πρέπει να μην γίνει ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Ανάταση χεριών. Λοιπόν, θα διαβάζω μόνο τους αριθμούς. Αρχίζουμε με την ε, πρώτη, την 5608. 5608 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 5609 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5610 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5611 και 12 είναι παρόμοιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 5613 και 14 α όχι με συγχωρείτε μόνο 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτω 14, 56, 15 και 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 56, 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 18 και 19 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 56-20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση υπέρ παρακαλώ και κρατήστε τα χέρια ψηλά να παραμείνουν ψηλά για να γίνει καταμέτρηση. Κατά. Ωραία, σαφέστερο το αποτέλεσμα. Αποχές απορρίπτεται. Επειδή δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα επαλήθευσης, να είσαστε σαφείς, σας παρακαλώ. 56-22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56-46 Συμβιβασμός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 23 και 24 καθώς και 25 καταπίπτουν. Η 26 έχει αποσυρθεί. 56-27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56.00, 28, 29 και 30 είναι παρόμοιες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 56.31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56.01. 32-33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 56-34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σαφώς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56-36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56.02 και 37 είναι παρεμφερής υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 56.05 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56.38 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να ξαναψηφίσουμε γιατί δεν ήταν απόλυτα σαφές το αποτέλεσμα. Υπέρ παρακαλώ να παραμείνουν τα χέρια ψηλά. Κατά. 22. Okay. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 κατά 18 υπέρ. 06 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-04 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5639 να με συγχωρείτε, κατά πίπτη και η 40, 5603 και 41 είναι παρεμφερείς, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται, 5647 είναι τροπολογία συμβασμού υπέρ, κατά, αποχές α, περνάει, 5642 πίπτη, εξαιτίας της τροπολογία συμβασμού, 43 υπέρ, κατά αποχές 5644 υπέρ κατά αποχές 5607 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5645 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά έχουμε και το σχέδιο γνωμοδότησης Στη συνέχεια τροπολογία 1 Βερζά. Ξεχωριστή ψηφοφορία ζητήθηκε από τους πρασίνους. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία συμβιβασμού 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 ή 4 καταπίπτει άρα πρέπει να ψηφίσουμε την 5 με μια προφορική. Από τον εισηγητή υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται. Όχι. Ψηφίζουμε την 5 με την προφορική του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 7 Κυρία Κέλλερ, θα ήθελα να προβάλλω μία προφορική στην ΕΠΤΑ. Να προσθέσουμε, ε, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα της στο Στοκχόλμης και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ιδιαίτερα με βάση τα νέα καθήκοντα όπως ορίζονται από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ωραία. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή τη μικρή προσθήκη. Όχι, ψηφίζουμε την 7 με την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ήθελα να το ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Ποιοι είναι υπέρ, ανάταση παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται με σαφήνεια 10. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 11, 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14, 14, δεν την ψηφίζουμε. 15, υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και Τώρα ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία. Φτάσαμε στην τελική. Α, μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Λειτουργεί τώρα το σύστημα. Και έτσι μπορούμε να δούμε όλοι πώς ψηφίσατε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται με πολύ μεγάλη ψηφοφορία, ε, πλειοψηφία με συγχωρείτε, 38 υπέρ, μία ε, ψήφος κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε με τις εργασίες μας. Σας παρακαλώ πολύ. Μετά την ψηφοφορία θα προχωρήσουμε στο εξή σημείο που είναι το 5. Μέτρα εφαρμογής της Συμφωνίας TFTP 2. Είναι ένα θέμα πληροφόρησης θα μας πληροφορήσει για τα μέτρα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα εφαρμοστεί δηλαδή το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας, FTP. Είχαμε ψηφίσει τον Ιούλιο επί του θέματος και στη συνέχεια όταν ο πρόεδρος Μπούζεκ έγραψε στον πρόεδρο Μπαρόζο για τα μέτρα αυτά, τα πρώτα μέτρα εφαρμογής, έγινε λόγος ε, για την, τον διορισμό ενός ε, εκπρόσωπου από, το Ευρωπαϊκό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του άρθρου 2 της Συμφωνίας και ζητήσαμε και το διορισμό ενός ανεξάρτου προσώπου για να εποπτεύσει τη διαδικασία διαχείρισης δεδομένων με βάση τη διαδικασία επαλήθευσης δυνάμει του άρθρου 4 και την κοινή ε, αναθεώρηση, όπως προβλέπετε. Πρόκειται για την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση, η οποία θα πρέπει να ισχύσει έξι μήνες μετά από τη θέση σε ισχύ της πρώτης συμφωνίας. Ο κύριος Ζωακίμ Νούνες Αλμέιδα θα μας ενημερώσει για το θέμα αυτό και για τις εξελίξεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την δυνατότητα να σας πληροφορήσω σήμερα για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας TFTP που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου. Κατανοούμε ότι θα θέλατε η συμφωνία αυτή να εφαρμοστεί όπου πώς προβλέπεται από, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα επί του θέματος. Θα ήθελα όμως να ζητήσω την κατανόησή σας, διότι ε, ορισμένα λειτουργικά καθαρά ζητήματα δεν μπορούν να συζητηθούν σε ένα ανοιχτό φόρουμ όπως ε, ισχύει στην παρούσα συνεδρίαση. Θα πρέπει να βασιστούμε στη, στην κοινοποίηση στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα εκεί όπου προβλέπετε και θα σας μιλήσω για την, τον διορισμό του επόπτη, τη διαδικασία ε, αναθεώρησης δυνάμει του άρθρου 13 και την εργασία της Europol για την εφαρμογή της συμφωνίας για να αρχίσουμε με τον ανεξάρτητο επόπτη. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά το διορισμό του ανεξάρτητου επόπτη, όπως ορίζεται από το άρθρο 12 της Συμφωνίας. Οι δραστηριότητες του, τα καθήκοντά του ή της, αφορούν την προσβασιμότητα στοιχείων από τη βάση δεδομένων TFTP θα πρέπει να αποκλείσει έρευνες αν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να γίνει έρευνα για συγκεκριμένα πρόσωπα, ο επόπτης ή επόπτρια θα πρέπει να δει κατά πόσο υπάρχει αιτιώδη συνάφεια σε σχέση με τις πληροφορίες που ζητούνται και τον σύνδεσμο με κάποια πτυχή της τρομοκρατίας. Όπως ορίζει το άρθρο 12, ο διοριστής ή η διοριστήσα θα πρέπει να ε, υπόκειται στην έγκριση από τις ΗΠΑ. Υπάρχει μία ανοιχτή θέση από τις 29 Ιουλίου και η προθεσμία υποβολής είναι η 15 Σεπτεμβρίου του 2010 η υποβολή αιτήσεων. Όταν λάβουμε τις αιτήσει, τότε θα προβούμε στην επιλογή. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα ενημερωθεί για την ε, εφαρμογή της, ε, του προγράμματος TFTP και σε σχέση με το διορισμό του ανεξάρτητου επόπτη καθώς και ως προς τους υποψηφίους και την τελική επιλογή. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, θα σας δώσουμε αυτές τις πληροφορίες ε, με βάση στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα που ορίζονται από τη Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ των οργάνων. Ο ανεξάρτητος, ένας ανεξάρτητος επόπτης έχει διοριστεί, αντίντεριμ, έως ότου πληρωθεί αυτή η θέση. Όπως ε, ανέφερε η Επίτροπος Μάνστρεμ, η διαδικασία έληξε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα ήθελα να σας αναφέρω, να αναφερθώ στο όνομα του επόπτη. Θεωρούμε ότι έχει την κατάλληλη πείρα έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και ο ενδιαφερόμενος εγκρίθηκε η υποψηφιότητά του, εγκρίθηκε από τις ΙΠΑ και ήδη έχει αρχίσει με τις εργασίες του, με τα καθηκοντά του. Έχετε πολλές ερωτήσεις ως προς τη συμφωνία στην αρχική της φάση και το διορισμό του ανεξάρτητου επόπτη. Ορισμένα ζητήματα ήδη έχουν υποβληθεί προς την Επίτροπο Μάλμστρεμ και θα λάβετε γραπτός απάντηση εν ευθέτω χρόνο. Ως προς τη διαδικασία αναθεώρησης, όπως γνωρίζετε, δυνάμει του άρθρου 13 προβλέπονται κοινέ αναθεωρήσεις και η πρώτη θα λάβει χώρα μετά από έξι μήνες, μετά δηλαδή από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Η αναθεώρηση αυτή θα λάβει υπόψη τα, το συνολικό χρηματοοικονομικό έλεγχο, τα κοινά στοιχεία μεταξύ Europol, Eurojust, κρατών μελών και τρίτων χωρών και θα δούμε πώς έχει χρησιμοποιηθεί οι, πώς έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές οι πληροφορίες για την πρόληψη ή αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και την προστασία δεδομένων όπως ορίζεται από τη Συμφωνία. Δυνάμη του άρθρου 13, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά την λήξη της αναθεώρησης αυτής. Γνωρίζετε ότι αυτή η διαδικασία αναθεώρησης ε, αφορά δύο αρχές προστασίας δεδομένων. Η μία θα προέρχεται από ένα κράτος μέλος, δηλαδή από εκεί όπου, από όπου προέρχεται ο επόπτης. Στις 5 ε, Αυγούστου λάβαμε επιστολή του κ. Γιάκοπ Κόνσταν που δουλεύει, που εργάστηκε με τις Ολλανδικές και Βελγικές αρχές ως προς την προστασία δεδομένων. Οι δύο αυτές αρχές θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αναθεώρησης. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες τον επόμενο μήνα και θα έρθουμε σε διαβούλευση μαζί σας πριν από την επόμενη διαβούλευση που προέρχεται με τις αρχές των ΙΠΑ. Έχετε ήδη υποβάλει ερωτήσεις τις οποίες, τις οποίες θα απαντήσουμε κατά τη διαδικασία αναθεώρησης και θα δοθούν απαντήσεις μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αναθεώρησης, για πρώτη τουλάχιστον φορά. Ως προς το ρόλο της Europol, μέχρι την 1η Αυγούστου η Europol είχε αναλάβει αυτά τα καθήκοντα μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που προβλεπόταν, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επαλήθευσης που χρειάζεται δυνάμει του άρθρου 4 της Συμφωνίας για τη Συμφωνία της 30ης Ιουλίου μεταξύ Κομισιών και Αρχών ε, των ΗΠΑ. Αυτές ε, οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν μια συγκεκριμένη μονάδα από τη Europol, τη διαδικασία επαλήθευσης, τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης, θέματα εμπιστευτικού χαρακτήρα και ασφάλειας, καθώς και αιτιολόγηση των αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 4. Το έγγραφο ε, θεωρείται εμπιστευτικό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμπίπτει στη διαδικασία ε, κοινοποίηση στοιχείων μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της Europol, μάλλον στη Europol ανατίθεται και η διαδικασία απαλλαγής. Επίσης, ε, η μονάδα 04 θα πρέπει να αντιμετωπίσει την παρακολούθηση και την χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας με βάση δεδομένα από τις ΗΠΑ και θα γίνει επαλήθευση και απόφαση από τη Europol δυνάμει του άρθρου 4 της συμφωνίας. Η νέα μονάδα 09 επίσης θα αναλάβει την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 και μία ανταλλαγή ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης δυνάμει του άρθρου 4 έτσι ώστε η Europol να έχει περισσότερες αρμοδιότητες και γνώσεις για να καταπολεμήσει την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Έτσι θα έχουμε μια καλύτερη κατανόηση και συνεννόηση με τις ΕΠΑ τη στιγμή που οι ΕΠΑ προβάλλουν αιτήματα. Επίσης, η Europol θα αναλάβει καθήκοντα σε έναν τομέα που ε, την απασχολεί ήδη. Επίσης προβλέπεται μία νέα διαδικασία ανάλυσης στη Europol έτσι ώστε δυνάμει του άρθρου 4 να ταξινομούνται τα αιτήματα που προέρχονται από τις ΗΠΑ. Οι ανταλλαγές απόψεων με τις ΗΠΑ δυνάμει των άρθρων 9 και 10 θα κατατάσσονται σε αυτή τη διαδικασία ανάλυσης. Ως προς τις αρχικές μας ε, εμπειρίες είχαμε ένα αίτημα από τη ΣΥΠΑ δυνάμει του άρθρου 4 της συμφωνίας στις αρχές Αυγούστου του 2010 και μετά την επαλήθευση της Europol δόθηκε άδεια. Επίσης, ο αρμόδιος ενημερώθηκε και σε επίπεδο νομικής υπηρεσίας και προστασίας τράπεζας δεδομένων της Τράπεζας Δεδομένων. Επίσης, δυνάμει του άρθρου 9 της Συμφωνίας δόθηκαν ορισμένα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και τα άρθρα 9 και 10 συμβαδίζουν με όλους τους όρους της συμφωνίας καθώς και τα αιτήματα που προέρχονται από τη ΣΥΠΑ και σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να σας δώσω επιχειρησιακά στοιχεία σε ένα ανοιχτό φόρουμ όπως το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νούνες Αλμέιδα. Νομίζω ότι ορισμένοι θα ήθελαν να υποβάλουν ερωτήσεις. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινώς έχω εκπλαγεί. Δεν ξέρω αν είναι και θετική έκπληξη αυτή για τα όσα είπε Αλμέιδα γιατί βλέπω ταχύτητα αντιδράσεων που δεν έχουμε συνηθίσει. Για να είμαι όμως βεβαία ότι κατανόησα καλά θα κάνω μια ερώτηση. Από διάφορες συνομιλίες που έχω διεξαγάγει γνωρίζω πόσο περίπλοκες είναι οι τεχνικές προϋποθέσεις και άλλα μέτρα για την λειτουργία για παράδειγμα της Ευρωπόλ. Παρόλη την περιπλοκότητα ωστόσο του θέματος αυτό που κατάλαβα είναι ότι από 1η Ογδόου είναι δυνατόν να διαβιβάζονται δεδομένα στις πρώτης Ευρωπόλ είναι πλήρως σε θέση να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κρίνει μια αίτηση και μόνο μετά από έγκρισή της Ευρωπόλ διαβιβάζονται τα δεδομένα. Επίσης έχω και μια ερώτηση σχετικά με τον ελεγκτή ο οποίος υποτίθεται ότι δραστηριοποιείται από πλευράς Αμερικανών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να συμμετάσχει. Η ερώτησή μου είναι εάν μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής προβλέπεται κάτι τέτοιο ή εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία θα κάνει αποκλειστικά την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν μεταξύ των προσώπων εκείνων που επιθυμούσαμε να υπάρξει μια λογική συμφωνία. Και δεν το μετανιώνω, όμως εκφράζω τώρα κάποιες ανησυχίες. Βλέποντας το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, μου προκαλείται ανησυχία σχετικά με την διαφάνεια της διαδικασίας και με τη συνέχισή της. Η Επίτροπος Βάλεφτρομ είπε ότι διορίστηκε επόπτης επί προσωρινής βάσεως. Μας είπατε τώρα ότι δεν μπορείτε να αποκαλύψετε το όνομά του. Από τον τρόπο που διατυπώσατε αντιλαμβάνομαι ότι είναι αρσενικού γένους. αλλά τέλο πάντων αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε να αποκαλύψετε το όνομα, γιατί άραγε να είναι απόρριτο το όνομα. Και αν αυτό είναι θέμα, τότε αυτό μου δείχνει ότι η υπόλοιπη διαδικασία δεν θα είναι διαφανής. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση, διότι ήταν δημόσια διαδικασία επιλογής. Είπατε και για την επιστολή του Πρόεδρου Μπούσεκ που ζήτησε συμμετοχή του Κοινοβουλίου και που υποτίθεται ότι θα μας υποβάλλονταν τα τρία ονόματα υποψηφίων και θα μπορούσαμε και εμείς να συμβάλλουμε με εκφράση άποψη για την επιλογή του επόπτου. Τώρα, πότε θεωρείτε ότι θα ολοκληρωθεί η δικασία επιλογής του υποψηφίου και μπορείτε να μας βεβαιώσετε ότι θα είναι διαφανής η διαδικασία και το κοινοβούλιο θα εμπλέκεται, ναι ή όχι. Αν θυμούμε καλά, και είμαι βεβαία ότι θυμούμε καλά, τούτο εδώ ήταν προϋπόθεση για την υπογραφή της συμφωνίας. Και διόλου δεν μας αρέσει να βλέπουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει σε λιγμούς για να το αποφύγει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αλβάρο νομίζω. Όχι. Όχι, καλά, φαίνεται, φαίνεται πως έκανα λάθος. Ωστόσο λαμβάνει το λόγο ο κύριος Άλβαρο. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, χάρη στα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου. Συμφωνώ με την κυρία Βέμπερ. Εμείς συνεργαστήκαμε καλά με τα αναθεσμικά όργανα και μάλιστα πράξαμε τα δέοντα πριν ακόμα να εκπληρωθούν τα υπεσχημένα από, από τα άλλα θεσμικά όργανα. Ίσως τώρα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Τώρα για την προσωρινή επιλογή, ίσως θα μπορούσε να έχει γίνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως την διαφάνεια της μελλοντική διαδικασίας, ε, εδώ μπορεί να παρέμβει διαφωτιστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε με κλειστά μάτια να επιλέξουμε κάποιον και να τον διορίσουμε. Είναι φυσικό να επιμένουμε ώστε, η Ευρωπαϊκή, ε, ώστε το πρόσωπο που θα επιλεγεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας και θα το κατανοήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω. Αλμπρεχτ Είναι κάπω σαν ε, θεωρία τη συνωμοσία να μιλούμε τώρα για την προστασία δεδομένων του προσώπου που θα είναι αρμόδιο για την προστασία δεδομένων. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει το πρόσωπο αυτό. Η μεγάλη νίκη λοιπόν που επιτύχαμε πριν από τι θερινέ διακοπέ ώστε να μην είναι και τόσο σημαντική τέλο πάντων. Πάντω τώρα έχω δύο σχόλια διότι βέβαια το άθο 12 αξιώνει διορισμό με πλήρη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της παρούσας Επιτροπής. Πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή ότι θα διοριστεί κάποιος που έχει τα εξή προσόντα κλπ. λοιπά. να γίνει τώρα προσπάθεια να ε, περιγραφεί αυτό εδώ βάζοντας προσωρινά κάποιον. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο σχόλια που επιθυμώ να κάνω. Πρώτο, ότι παρακαλέσαμε τον πρόεδρο Μπούσεκ να αρχίσει διάλογο με το Κογκρέσο σχετικά με την προστασία δεδομένων που διαβιβάζονται υπερατλαντικά. Θα είναι σωστό νομίζω να τον ρωτήσουμε αν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Και το δεύτερο για το TFTP είναι σχετικά με την Ευρωπόλ. Εδώ δεν είναι ερώτηση προς την Κομισιόν, αλλά ερώτημα που το, θέτω για μας. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να ρωτήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει είναι και σύμφωνοι με τη συνθήκη, αν έχουμε δώσει τον εποπτικό ρόλο δηλαδή στην Ευρωπόλ. Εμείς ως πράσινοι ρωτήσαμε και πριν από τις θερινές διακοπές και μας απαντήσανε τότε ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, είμαστε νομοθέτες κτλ. Εγώ νομίζω όμως ότι είναι καλή ιδέα να ρωτήσουμε τώρα εάν αυτά τα συστήματα διαβιβάσεως που περιλήφθηκαν στη συμφωνία TFTP συμβατίζουν με τις διατάξεις της νέας συνθήκης. Και θα, θα χαιρόμουν πολύ εάν μπορούσε να συμφωνήσει η πλειοψηφία της παρούσας Επιτροπής να θέσει το ερώτημα στην Επιδυνομική Επιτροπή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία Ένστ. Ευχαριστώ. Εγώ εκφράζω την κατάπληξή μου. Μέχρι την έναρξη των θεσμών διακοπών λέγαμε ότι όλα θα πρέπει να είναι διαφανή, θα πρέπει να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Μας δόθηκε αυτή η διασφάλιση εκατοντάκης και τώρα τα βλέπω όλα απόρριτα. Μα από ποια στιγμή και μετά ισχύει ο εμπιστευτικό χαρακτήρας, ποια πράγματα είναι απόρριτα και ποια όχι. Και για μας τι σημαίνει, θα έχουμε και άλλες τέτοιες παρουσιάσεις όπως τώρα που θα μας λένε δηλαδή ότι εδώ σε ανοιχτό δημόσιο κύκλο δεν μπορούμε να τα πούμε. Ε, τότε πότε θα τα πούμε. Θα πάμε να τα πούμε στο καφενείο ξεχωριστά, σε πηγαδάκι, εμείς οι βουλευτές. Αυτή λοιπόν η τήρηση απόρριτου μου φαίνεται ότι δεν είναι αρμόζουσα εν προκειμένου. Και δεύτερη ερώτηση τώρα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πώς συμπεραίνεται ότι είναι απόλυτα προετοιμασμένη η Ευρωπόλη για να λάβει το ρόλο αυτό και ήδη από πρώτης ογδόου ξεκίνησε και αναλαμβάνει και καταφέρνει και κινεί και τα λοιπά. Τι πάει να πει η Ευρωπόλ ήταν από την αρχή σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά με επιτυχή τρόπο ήδη από πρώτης ογδόου. Θα ήθελα να μου πείτε λίγα περισσότερα εν προκειμένου. Ευχαριστώ. Εγώ βλέπω τα πράγματα λίγο πιο θετικά από τους προηγούμενους. Το λέω διπλωματικά. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα πολλά έχουν επιτευχθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τότε δηλαδή που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που μας ενημέρωσε για το τι συνέβη σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα και επίσης θεωρώ ικανοποιητικό το ότι έχουν γίνει πολλά ήδη. Δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει όλα ή ότι θα έπρεπε να είμαστε πλήρω ικανοποιημένοι. Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πολλά πράγματα έχουν ήδη γίνει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο σχολείο μου είναι το εξή. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να σεβαστούμε δηλαδή τις αρμοδιότητες του κάθε οργάνου. Ο δικός μας ρόλος είναι σαφής και θα πρέπει να ελέγξουμε προσεκτικά το έργο της Κομισιόν. Έτσι θεωρώ, αυτό θεωρώ, αυτός θεωρώ μάλλον ότι είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου και ε, θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε με ζήλο. Δεν θα πρέπει όμως να σφετεριστούμε αρμοδιότητες οι οποίες και δικαίως και υπό την συμφωνία αυτή ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να υπερβούμε τι αρμοδιότητά μα γιατί τότε θα προκύψει σύγχυση. Α γίνουν τα πράγματα λοιπόν όπω πρέπει, ας αφήσουμε την Κομισιόν να πράξει τα όσα εμπίπτουν στι αρμοδιότητε τη και μετά α συζητήσουμε και α διαμορφώσουμε πολιτική κρίση στην βάση των πληροφοριών που θα μα θέτει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν λέω ότι θα συμφωνούμε πάντοτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράγματι, στο παρελθόν διαφωνήσαμε και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες όπου θα διαφωνήσουμε. Όμως, <clears throat> ας σεβαστούμε τον ρόλο που της αναθέτει η συμφωνία. Μπρόνς. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μπορεί να μας πει ή να μας θυμίσει εάν υπό την τελική μορφή της συμφωνίας θα μπορούν οι Ηνωμένε Πολιτείε να διαβιβάζουν δεδομένα που λαμβάνουν από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες χώρες τρίτες και κυρίως συμμάχους τους στην ε, Έγκυς Ανατολή που θα τους επιτρέπει ε, που θα τους επιτρέψει ίσως τις χώρες αυτές να προβούν σε παράνομες πράξεις όπως η πρόσφατη δολοφονία στο Ντουμπάι. Ευχαριστώ. Κυρία Ιντφέλτ. Εγώ θα συμφωνήσω με τα λεχθέντα πολλών εκ των συναδέλφων μου. Και εγώ παραμένω έκπληκτη και απογοητευμένη από τον μυστικό χαρακτήρα των δρο, δρομένων από την Κομισιόν. Ναι κύριε Πουσουτήλ, να συμφωνούμε, να σεβόμαστε μάλλον τον ρόλο της Κομισιόν, αλλά να σεβόμαστε όμως και τα δικαιώματα των πολιτών. Έχει ευθύνε και απέναντι στους πολίτες, δηλαδή μέγιστη διαφάνεια. Μέγιστη διαφάνεια. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στην προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαβιβάζει τραπεζικά δεδομένα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών στους Αμερικανούς χωρίς καμία εγγύηση, καμία εξασφάλιση, ενώ ταυτόχρονα να καλύπτει με τον μανδύα της εμπιστευτικότητας το όνομα του επόπτη. Αντιστρέφει τα πράγματα. Τα αναποδογυρίζει. Έχουμε δικαίωμα να μάθουμε ποιο θα είναι το πρόσωπο αυτό και να ελέγξουμε την διεξαγωγή της διαδικασίας. Και κάτι άλλο. Τίθεται και θέμα εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων η Κομισιόν γνωρίζει καλά τη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε για να περάσουμε την συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Και πολλοί την υπερψηφίσαμε τελικά με πολλέ επιφυλάξει. Εν πάση περιπτώσει, επαφεθήκαμε σε μια εμπιστοσύνη. Δεν είμαι βέβαια τώρα ότι προέβαινε στη σωστή επιλογή. Αναμένω, εάν εμπιστεύομαι την Κομισιόν, η Κομισιόν να κάνει πάντο το δυνατό για να κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτή. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά και για άλλε μελλοντικέ. Και αν δεν έχουμε, αν δεν μπορούμε να σας εμπιστευτούμε τυφλά, τότε όλα θα πρέπει να τα κάνουμε γραπτός μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Και κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι μπορεί να τελεσφορήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αποβεί αξιόπιστος εταίρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ας αρχίσει από τη διαφάνεια. Ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπλήσωμαι τώρα που μόλις άρχισε η δουλειά και ε, έχουμε κατακλείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τώρα με καχυποψία. Εντάξει, και εγώ είμαι ιδιαίτερα επικριτική σε αυτή τη συμφωνία, αλλά προσπαθεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει αυτά που εμείς αποφασίσαμε στο Κοινοβούλιο και χαίρομαι που με μεγάλη συνέπεια από ό,τι φαίνεται το πράττει. Αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω και τη μεγάλη μυστικοπάθεια πουθενά. Και λέω ως βουλευτής ότι δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση εγώ να επιλέξω ποια πρόσωπα είναι ε, τα πλέον ενδεδειγμένα και έχουν τα προσόντα για να είναι υπόπτες. Ε, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επιλέξει τους καλύτερους ειδικού με τα αντίστοιχα προσόντα. Αυτό δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των κομμάτων. Και θα ρωτούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποιου όρου και προποθέσει θα μπορούσαμε να μάθουμε αυτό το όνομα. Γιατί εντάξει και το όνομα ας πούμε τι θα πούμε, τι θα ξέρουμε, το ξέρουμε. Αν είναι ο κατάλληλο, ο καταλληλότερο άνθρωπος, ο αρμοδιότητα, στον βαθμό που γνωρίζω την ε, Europol και ε, τους θεσμούς, οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί είναι πραγματικά ειδικοί στου τομεί του και σίγουρα θα έχουν βρει κάποιον μια προσωπικότητα που θα είναι ακριβώς ο ειδικό σε αυτά τα θέματα. Ας μην ασκούμε τώρα και μάλιστα με πληθώρα ε, την προληπτική κάχη υποψία. Ας περιμένουμε όπω είπε και ο Σάιμον Πούσου, λιγου μήνε να δούμε ε, πώς θα έχουν επεξεργαστεί τα θέματα αυτά και ποιε είναι οι γνωμοθετήσεις και τότε θα αποφανθούμε. Τώρα άρχισε η δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε καν να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για ε, την εργασία. Μόλις ε, δόθηκε το ενακτήριο λάκτισμα, και εγώ έτσι κατάλαβα την έκθεση αυτή. Δεν θεωρώ ότι είναι μια έκθεση συνολική ε, που μας ενημερώνει για τα πάντα, τι σχεδιάζεται, ποιες διαδικασίες ισχύουν και ποιο και υποθέσεις. Καταλαβαίνω αυτά που ρωτάτε για την προστασία των δεδομένων. Κύριε Άμπρεχτ, εσείς είστε ειδικό. Η προστασία των δεδομένων δεν αφορά μόνο τον εαυτό μας. Ενδιαφέρει και κάποιες αρχές που εργάζονται σε πάρα πολύ ευαίσθητα ε, χωράφια, όπως είναι ας πούμε, ο τομέας της τρομοκρατίας. Για αυτούς δεν ισχύει πια η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουν και εκείνοι το δικαίωμα. Και κανονικά εμεί δεν συνεδριάζουμε στα καφενεία των βουλευτών, αλλά συνεδριάζουμε και κλεισμένων των θυρών όταν είναι τα θέματα εμπιστευτικά ή απόρριτα. Και αν θέλετε να φέρω και καφέ και γλυκό για τις συνεδρίες και κλεισμένων των θυρών, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Mr. Mello. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα για πληροφόρηση καθαρά. Δηλαδή το πρόσωπο για το οποίο μιλάμε είναι το ίδιο με το οποίο με αυτό που αναγράφεται σε αυτό το έγγραφο σε σχέση με το προσωρινό προσωπικό. Είναι, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Όχι, μιλάμε για το θέμα που αφορά την ημερήσια διάταξη, δηλαδή για την παρακολούθηση πληροφορίας σε σχέση με τον διορισμό του προσώπου αυτού για την παρακολούθηση και τον οικονομικό εντοπισμό. δηλαδή για την αναθεώρηση και τα δεδομένα όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της συμφωνίας που εγκρίθηκε τον Ιούλιο. Να, αλλά νομίζω ότι μόνο σε αυτό το στοιχείο αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο και αν πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, νομίζω τότε αυτό σημαίνει ότι προτρέχουμε, γιατί αυτό το έγγραφο, στην πρώτη τελευταία παράγραφο, λέει ότι η προθεσμία είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2010 για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Πώς μπορεί να έχουν επιλέξει, να έχει γίνει επιλογή του προσώπου τη στιγμή που δεν έχουν υποβληθεί όλες οι υποψηφιότητες. Αυτό είναι παράλογο. Δεν θα ήταν σκόπιμο να περιμένουμε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 και με βάση τις υποψηφιότητες να ξέρουμε ποιος θα επιλεγεί. Γιατί εδώ υπάρχουν συνάδελφοι που ε, ρωτούν ποιος ε, επελέγει χωρίς να έχει λήξει η διαδικασία. Γι' αυτό μου φαίνεται παράλογο διότι με βάση, τις, ε, με βάση αυτά που αναφέρθηκαν φαίνεται το πρόσωπο είναι το ίδιο με αυτό που αναγράφεται εδώ. Μιλάμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι η ΕΠΑ είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, δεν είναι εχθρή μας. Και βλέπω να υπάρχει μία αμφισβήτηση των είπα μία δυστημία γενικότερα. Διότι πρόκειται για μία δημοκρατική χώρα, καταπολεμεί την τρομοκρατία και είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος. Κατανοώ τις ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις βασικές ελευθερίες. Νομίζω ότι δεν μπορεί ο οποιοδήποτε βουλευτής να θεωρεί ότι καταπατώνται δικαιώματα και βασικές ελευθερίες. Γιατί οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στη ΣΥΠΑ είναι οι ίδιες πληροφορίες που έχουμε και εμείς σε σχέση με τρομοκρατικές δράσεις. Γιατί όταν υπάρχει κάποια τρομοκρατική ενέργεια στις ΗΠΑ κοινοποιείται στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΗΠΑ είναι λοιπόν ο βασικός μας σύμμαχος, είναι μια δημοκρατική χώρα, υπερασπίζεται τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες και αξίες και υπ' αυτή την έννοια ε, συμμεριζόμαστε τις ίδιες αρχές. Άρα μιλάμε για διαφάνεια δικαιωμάτων, ελευθεριών και εγγύσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε μία κοινή προσπάθεια, κάτι το οποίο δεν γίνεται μέχρι τούδε. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, παραχωρήθηκαν πολλά, τα οποία δεν είχαν παραχωρηθεί στο παρελθόν. Υπάρχουν επιφυλάξεις. Εγώ όμως είμαι ε, ε, ριζοσπαστικός δημοκράτης. Όμως σε θέματα τρομοκρατίας δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ε, μία επιμερισμένη, μία διαφορετική διαλεκτική. Δεν μπορούμε παρά να κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες διαφορετικά. Η επιφύλαξη αυτή θα ήταν εντελώς αντιπαραγωγική. Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από όλα τα θεσμικά όργανα. Έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 να μην αποφανθούμε, διότι τότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος υποψηφιωτήτων και τότε θα γίνει και η τελική επιλογή. Γι' αυτό τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν, δηλαδή το όνομα του προσώπου, μάλλον είναι ένα μεγάλο λάθος. Το... Συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Μέλο. Ε, να σας θυμίσω ε, το σημείο της ημερήσιας διάταξης που ορίζει ότι είναι τα πρώτα μέτρα εφαρμογής συμφωνίας για το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Γι' αυτό μας ενημερώνει η κυρία ε, ο κύριος, συγγνώμη, πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι κυκλοφόρησε και η προσωρινή ε, θέση που προκηρύχθηκε για τον επόπτη, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για τη διαχείριση των κρίσεων κτλ. Στην προκήρυξη που αναφέρθηκε ο κύριος Μέλλο, ε, χρειάζεται ενδεχομένω ε, διευκρίνηση. Ε, θα το επαληθεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα έχει ανοίξει η συζήτηση, έχουν ζητήσει πολλοί συνάδελφοι το λόγο, αλλά να περιορίσουμε το χρόνο αγόρευσης, γιατί δεν θα προλάβουμε. Γιατί έχουμε προσθέσει και άλλο θέμα στη συνεδρίαση των συντονιστών και θα χρειαστεί χρόνο. Έχει προσκληθεί και η νέα Γενική Διευθύντρια Δικαιοσύνης, η κυρία Λεβάη να συμμετέχει και επειδή θα τελειώσουμε στις 6.30 αλλιώς κάθε λεπτό που θα περνάει μετά τις 6.30 θα πρέπει να ζητάμε συγγνώμη από τους διερμηνείς μας. Κύριο Σταβάρης. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Νομίζω ότι αρχίσαμε πολύ άσχημα. Είναι μια πολύ κακή αρχή. Υπάρχουν ε, ε αντικρουόμενες πληροφορίες και από όσο γνωρίζω, οι πληροφορίες της Κομισιόν πέρασαν και στον τύπο. Άρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς τη διαδικασία διαφάνειας όπως μας είχε υποσχεθεί η Επιτροπή στην περίπτωση του SWIFT. Είχαμε τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Στιουαρτ Λεβι στις 11 Ιουλίου όπου και αναφέρθηκε τα δεδομένα αυτά στην Guardian ότι το SWIFT ήδη πιάνει τρομοκράτες. Αυτό ε, τυπώθηκε, μάλλον αναφέρθηκε στον τύπο λίγο μετά την 11η Ιουλίου. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή τι κάνει το SWIFT, ήδη πιάνει τρομοκράτες, σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Σε σχέση τώρα με τον ε, διορισμό του επόπτη, του Ευρωπαίου επόπτη, στο TFTP, το γεγονός του ότι δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο αντίντεριμ ε, διοριστής δεν υπόσχεται τίποτα θετικό για το μέλλον, διότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε μαζί με το SWIFT και μια τροπολογία η οποία ακριβώς ανέφερε ότι θα πρέπει όλα αυτά να υπόκεινται στον έλεγχο και εποπτεία του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή μας ήταν πάντα πολύ ανοιχτή. Μπορούμε βεβαίως να συνεδριάσουμε και, και κλεισμένων των θυρών, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτή την πληροφορία. Ποιος έστω διορίστηκε αντίντεριν δεν μπορεί να μας αποκρύπτεται αυτή την ε, πληροφορία. Ίσως ο συνάδελφος έφτασε κάπως ε, αργά στην ε, Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, για την εφαρμογή του SWIFT θα πρέπει να υπάρχει μια σειρά εγγυήσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εδόθησαν διαχρονικά. Και εάν δεν εφαρμοστεί σωστά το SWIFT, τότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποσυρθεί και από το PNR, τα στοιχεία επιβατών δηλαδή, τη διαβίβαση δεδομένων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ύψος των περιστάσεων και δεν μπορεί να μας εγγυηθεί κανενός είδους διαφάνεια. Καλώς. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λούνε Σταλμέιδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω κύριε Λούνε Σταλμέιδα. Ε, για να τηρηθεί το απόρριτο που αφορά ορισμένα στοιχεία της πληροφορίας που θα περίμενε κανείς να μοιραστείτε με τα μέλη της Επιτροπής υπάρχει τεχνική διαδικασία σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας μας. Ε, δηλαδή είστε προσκεκλημένος να ε, παρευρεθείτε σε κεκλεισμένο το θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής μας για να ερώσετε τα μέλη της Επιτροπής. Και θα πρότεινα να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας αυτή και να έρθετε την επόμενη φορά το συντομότερο που θα συνεδριάσουμε και κλεισμένα των θυρών. Αμέσως μετά τη σύνοδο μιλήσει στο Στρασβούργο της άλλης εβδομάδας. Δηλαδή, στην επόμενη τακτική μας συνεδρίαση που θα είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή αλλά ήδη είχα προσφερθεί για κάτι τέτοιο και αυτό θα ήθελα ακριβώς να τονίσω. Δεν είπα ότι δεν θέλουμε να σας δώσουμε το όνομα του επόπτη, είτε είναι προσωρινός είτε είναι ο διοριστής αλλά δεν ήταν σκόπο να γίνει μέσα στα πλαίσια της παρούσης συνεδρίασης. Εμείς μπορούμε να σας αποκαλύψουμε το όνομα στο κατάλληλο φόρουμ μέσα στα πλαίσια πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα. Αυτά θα ήθελα να πω, αυτό θα ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Ωραία λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ λίγη αυτό το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσα υπάρχουν επιπρόσθετα σχόλια τα βάρες. Θα ήθελα μία διασάφηση. Σε σχέση με τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Σιουαρτ Λίβι σε σχέση με τα λεγόμενά του την 11η Ιουλίου. Τα στοιχεία άρχισαν να χορηγούνται μετά την 1η Αυγούστου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι έγινε μεταξύ 11η Ιουλίου και 1ης Αυγούστου που διέρευσαν αυτά τα στοιχεία δηλαδή από τον Υφυπουργό. Ε, κύριε Νούνες. δεν ε, βρίσκομαι στη δούλεψη του Υφυπουργού Λέβη. Άρα δεν είμαι υποχρεωμένος να σας πω γιατί είπε ή δεν είπε το οτιδήποτε, αλλά το πρόγραμμα ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια. Ο κύριος Λέβη αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το πρόγραμμα TFTP δεν άρχισε τώρα. Απλώς έχει τώρα την παρούσα μορφή, αλλά ίσχυε εκ των προτέρων. Άρα ο Υφυπουργό μιλούσε για δεδομένα τι ευτυπή πριν από την 1η Αυγούστου του 2010, όπου υπήρχαν μονομερείς ε, και συμφωνίες και διμερείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δύο-τρία χρόνια. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, αλλά μου φαίνεται λογικό, μου φαίνονται απόλυτα λογικές οι δηλώσεις του, γιατί προϋπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Τα βάρες. Άρα από την 11η Ιουλίου, από τις αρχές του Ιουλίου, τα στοιχεία, δικά μας στοιχεία δεν είχαν αποσταλεί στη ΣΥΠΑ. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Yes. Not on the basis of... Ναι, όχι με βάση τη νέα συμφωνία δεν είχαν διαβιβαστεί στοιχεία με βάση τη νέα σύμφωνη. Yes, we all understand Το ναι σημαίνει όχι. Ότι δεν είχαν διαβιβαστεί. Δεν είχαν διαβιβαστεί στοιχεία μέχρι την 1η Αυγούστου διότι δεν ίσχυε η συμφωνία. Άρα στην επόμενη ε, συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ θα μας δοθούν αυτές οι πληροφορίες από την Κομισιόν και κλεισμένων των θυρών. Στις 26-27 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων θα πρέπει να ε, διαθέτουν θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και ποιοι είναι οι υπήκοοι που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Η κυρία Τάνια Φαγιόν είναι η αρμόδια και θα θέλαμε να μας μιλήσει η Επιτροπή για τις αποστολές αυτές του καλοκαιριού κυρία Μπούς εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας πει πώς ε, έλαβαν, πώς έγιναν αυτές οι αξιολογήσεις στις δύο χώρες, στη Βοσνία, Ζεγοβίνη και την Αλβανία το καλοκαίρι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών για αυτό το θέμα είναι η αυριανή ημέρα. Αύριο την Παρασκευή λίγη η προθεσμία αύριο 3 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Και η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη συνεδρίασή μας, στις 13 Σεπτεμβρίου δηλαδή, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να ψηφίσουμε κατά τη δεύτερη ολομέλεια του Στρασβούργου. Κύριε Μπούς, έχετε το λόγο. Thank you, Um... Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, στις 27 Μαΐου 2010 η Επιτροπή ζήτησε απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ορίσαμε έναν αριθμό οροσίμων και όρων για αυτές τις χώρες όπου χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση. Και σας υποσχεθήκαμε να σας ε, μιλήσουμε για τα αποτελέσματα αυτών των αποστολών που έγιναν τον Ιούλιο στη Βοσνία Αρζεγοβίνη από τις 5 μέχρι τις 8 Ιουλίου και στην Αλβανία από τις 12 μέχρι τις 15 Ιουλίου. Η έκθεση που προπαρασκευάζει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή βασίζεται στις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που συμμετείχαν στις αποστολές σε άλλες πηγές της Επιτροπής καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία που λάβαμε από τις χώρες κατά τα τέλη Ιουνίου και Αυγούστου. Με βάση αυτά τα στοιχεία βρισκόμαστε στην τελική μορφή της αξιολόγησης θα αξιολογήσουμε τα υπολοιπόμενα κριτήρια για την Αλβανία και τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Θα έχετε ένα έγγραφο εργασίας το, στο οποίο θα δοθεί τελική μορφή κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Άρα μπορώ να σας δώσω μόνο ορισμένα προκαταρκτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτών των δύο αποστολών σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές της Αλβανίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αρχίζοντας από την Αλβανία λοιπόν και σε σχέση με τον ορισμό μιας στρατηγικής για να ορίσουμε την επανεισδοχή των παλινοστούντων στην Αλβανία υπάρχει μια ε, στρατηγική για την περίοδο 2010-2015 για τους ε, παλινοστούντες εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2010 και υπάρχει ένας εκτενής ε, μηχανισμός για την ένταξη των ε, παλινοστούντων. Το πρόγραμμα δράσης και η στρατηγική αφορούν τις βασικές ανάγκες των παλινοστούντων όπως η εγγραφή στα Μητρώα, στέγη, εκπαίδευση και απασχόληση. Καταβάλλονται προσπάθειες για την ε, πραγματική εφαρμογή του προγράμματος δράσης και της στρατηγικής ως προς την ε, εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, οι αλβανικές αρχές επιτελούν τη σωστή, τη σωστή πρόοδο. Ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, ανοιχνεύουμε τις προσπάθειες αυτές μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας και με τις ανακριτικές αρχές. Ε, αρχές που παρακολουθούν την εφαρμογή του ε, νόμου έχουν ενισχυθεί και υπάρχει συνεργασία μεταξύ αρχών ε, που ελέγχουν την επιβολή του νόμου καθώς και ανακριτικές και αστυνομικές αρχές. Είναι ε, είναι ευκταία περαιτέρω βήματα προόδου έτσι ώστε να έχουμε και μια σωστή αποτίμηση κινδύνου. Ως προς την, ε, τις ανακριτικές διαδικασίες και τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος υπάρχουν κοινέ ε, ομάδες συνεργασίας και βλέπουμε μια αύξηση, μια καλύτερη μάλλον αντιμετώπιση παρομοίων θεμάτων. Θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, δηλαδή να είναι πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση του αργωνωμένου εγκλήματος. Ως προς το τρίτο ορόσημο έχει επιτελεστεί πρόοδο σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου σε σχέση με την κατάσχεση εμπορευμάτων και αγαθών μέσα στα πλαίσια του οργανωμένου εγκλήματος και των περιουσιακών στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος, έτσι ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος σε σχέση με την κατάσχεση περιουσιακών δεδομένων που απορρέουν από το έγκλημα. Γίνεται κατάρτιση του προσωπικού για να μπορέσουν να ειχνηλατήσουν τα παράνομα αυτά περιουσιακά στοιχεία. Και αυτό αφορά και μία ειδική μονάδα ε, πληροφόρησης ως προς τα οικονομικά στοιχεία και την εφαρμογή του νόμου. Η ευρωστία του νέου νόμου δοκιμάστηκε ε, ενώπιον του Αλβανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που θα αποφανθεί ως προς την συνταγματικότητα του νόμου την επόμενη εβδομάδα. Σε σχέση με τα τρία ορόσημα για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την ενίσχυση των δυνατοτήτων και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, οι αρχές επιτελούν μια πολύ καλή πρόοδο και ως προς την εφαρμογή της νομικής βάσης και το πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση του εγκλήματος έχει επιτελεστεί πρόοδος, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση του χρηματικού του οικονομικού εγκλήματος και επίσης οι διοικητικέ ε, αρχές ακολουθούν ε, στοχοτατημένες ενέργειες και κατάρτιση έτσι ώστε να υπάρχουν και τα επαρκή χρηματοδοτικά μέσα αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης η συνεργασία έχει ενισχυθεί όπως δείχνουν ορισμένες επιτυχείς δράσεις. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, διαγράφεται μια πολύ καλή τάση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε, σε μια φάση δίωξης και ανάκρισης, ανακριτικής διαδικασίας για ορισμένες ε, πολύ σοβαρές υποθέσεις, καθώς και για υποθέσεις ελάσσονος σημασίας. Θα πρέπει να καταρτιστεί μια νέα υπηρεσία κατά πολέμηση της διαφθοράς. Ως προς τα ηλεκτρονικά στοιχεία και το πρόγραμμα δράσης και τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ διοκτικών αρχών και αστυνομικών αρχών υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και οι αρχές εφαρμογής του νόμου και ελέγχου εφαρμογής του νόμου συνεχίζουν αυτή τη συνεργασία έτσι ώστε να αναβαθμιστούν αυτές οι δυνατότητες. Υπάρχει μια ειδική ε, μονάδα σε επίπεδο αστυνομικών αρχών για ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, έχει συσταθεί αυτή η αρχή, έχει επανδρωθεί και υπάρχουν και τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα. Επίσης έχει εγκριθεί το οργανόγραμμα του οργανισμού αυτού ως προς την ε, εθνική οργάνωση και την εφαρμογή του, του ποινικού δικαίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και το όλο πλαίσιο ε, μετά από διαχείριση, από εξέταση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο εγκρίθηκε τον Αύγουστο. Πρόκειται για, μια, για προκαταρκτικά στοιχεία που σας δίνω, αλλά τα στοιχεία είναι αρκετά θετικά ως προς τις πληροφορίες που λάβαμε από τις εθνικές αρχές. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι επιτελέστηκε μεγάλη πρόοδος από το Μάιο του 2010 και τα δύο κράτη μπορούν να ανταποκριθούν. Θα θέλαμε να τις ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν αυτή την πορεία μέχρι την πλήρη έγκριση όλων αυτών των οριοθετήσεων, οροσίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κοινοποιήσει την έκθεση στο Κοινοβούλιο και Συμβούλιο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν για την έγκριση, για την ενδεχόμενη έγκριση της πρότασης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λέει και ο Πρόεδρος. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε από την εισηγήτρια. Θα θέλατε το λόγο, η κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι διότι σήμερα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές μας δίνει τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις, μετά τις αποστολές αξιολόγησης δεδομένων στην Αλβανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έχουμε περισσότερους ενδιαφερόμενους εδώ από ό,τι βλέπω σε σχέση με τη συνεδρίασή μας ε, του Ιουλίου και πολλοί παρακολουθούν την ε, εξέλιξη της διαδικασίας. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι διότι έχει επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος και στις ε, δύο χώρες. Είμαι πεπισμένη ότι οι αντίστοιχες κυβερνήσεις ε, το τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες επένδυσαν πολύ σε αυτή τη διαδικασία απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων. Άρα, είπατε ότι θα μας δώσετε μάλλον τα τελικά στοιχεία σε δύο εβδομάδες. Από ό,τι βλέπω όλη η προεργασία είναι πολύ θετική και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση. Ε, για μια τεχνική καθαρά διαδικασία και έτσι θα πρέπει να παραμείνει μέχρι τέλους. Υπάρχει ίση μεταχείριση με όλες τις χώρες της Δυτικών Βαλκανίων, Σερβία, Μακεδονία και Μαυροβούνιο γιατί αυτό ακριβώς το καθεστώς ακολουθήσαμε και μέχρι το Δεκέμβριο για εκείνες τις χώρες. Βρισκόμαστε ε, ένα χρόνο μετά και υπάρχουν άλλες δύο υποψήφιες χώρες που θέλουν να απαλλαγούν από αυτό το υποχρεωτικό καθεστώς θεωρήσεων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο στοιχεία. Τον Ιούνιο, πέρσι τον Ιούνιο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία νομοθετική πρόταση για, τρίτες, για τρεις χώρες. Ήδη ξέραμε την ημερομηνία απελευθέρωσης. Είχαμε μιλήσει για την 1η Πρώτου 2010. Ε, έγινε και πριν πριν από τα Χριστούγεννα. Σήμερα δεν ξέρουμε τις ημερομηνίε για την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μετά από την ομοθετική δηλαδή πρόταση της Επιτροπής. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ίση μεταχείριση. Θα πρέπει να μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και να κρατήσουμε την υπόσχεσή μας. Πέρσι τον Νοέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε με κοινή δήλωση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την υπόθεση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και Αλβανίας όταν ανταποκριθούν στα κριτήρια. Και είπαμε ότι θα το κάνουμε αυτό επιγόντως. Τη στιγμή που πληρούνται οι τεχνικοί όροι, δεν έχουμε κανένα λόγο για περαιτέρω καθυστερήσεις. Ε, ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει απελευθέρωση του καθεστώτος ε, θεώρησης. Και στην εκστρατεία μας ε, μιλήσαμε για ε, ελεύθερη κυκλοφορία, το οποίο δεν σημαίνει αναζήτηση θέσεων εργασίας ή αναζήτηση ασύλου το θέμα αυτό επιλήθηκε και με τις ε, τρεις προγενέστερες χώρες. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εκστρατεία, μιλάμε για ελεύθερη κυκλοφορία μέχρι 90 ημέρες. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί και θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση τέλος. Να συνεχίσουμε να πιέσουμε, να ασκήσουμε πίεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, έχουμε μία συγκεκριμένη στενή προθεσμία και γι' αυτό είναι δική μας ευθύνη να φέρουμε αυτή τη διαδικασία στο τέλος της. Μας έδειξαν εμπιστοσύνη, δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. και θα πρέπει να μας απασχολήσει και το κοσυφοπέδιο στο εγγύς μέλλον. Δεν πρέπει να, το, να αφήσουμε αυτό το, το μεγάλο κενό ε, σε σχέση με την όλη κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουζούτη έχει το λόγο. Τον ζητήσατε. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Well, let me on behalf of the EPP group also extend... Θα ήθελα εξ ονόματος του ΕΛΚ να εκφράσω τη θέλησή μου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην Αλβανία και Βοσνία Αρζεγοβίνη με μεγάλη μας χαρά, δηλαδή θα πρέπει να επιτελέσουμε το δικό μας σκέλος της εργασίας για να βοηθήσουμε τους φίλους σε αυτές τις δύο χώρες για να μπορέσουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και το δικό τους σπίτι, όπως είναι και το δικό μας. Συμφωνώ με την Τάνια Φαγιόν και θα ήθελα να τη συγχαρώ για την εργασία της ε, επί του θέματος αυτού. Η θέση του ΕΛΚ ήταν ότι εφόσον πληρούνται οι τεχνικοί όροι, τότε θα πρέπει να υποστηρίξουμε την απελευθέρωση θεωρήσεων για αυτές τις δύο χώρες, όπως ακριβώς κάναμε και με άλλες χώρες των Βαλκανίων πέρσι. Αναμένουμε δηλαδή με θέρμη τα αποτελέσματα της πλήρωσης αυτών των απαιτήσεων. Πιστεύουμε ότι θα είναι θετική η έκβαση και εμείς θα τηρήσουμε το λόγο μας ως προς την απελευθέρωση των θεωρήσεων το ταχύτερο δυνατόν. Άρα το ΕΛΚ θα συμφωνήσει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Φαγιόν που παρακολούθησε αυτή την διαδικασία με ακρίβεια και με αφοσίωση. Έχετε απόλυτο δίκιο, πέρασε ένας χρόνος από τότε που οι Σέρβοι έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συζητήσαμε τότε μεταξύ μας και είπαμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια ή διαδικασία για την Βοσνία Ζεγοβίνη και την Αλβανία, τη στιγμή που πληρούνται τα κριτήρια και τη στιγμή που ισχύει κάτι τέτοιο, από ό,τι φαίνεται, που μάλλον θα ισχύσει, τη στιγμή δηλαδή που πληρούνται τα κριτήρια, ε, η ώρα και θα πρέπει να έχουν αυτή την ελευθερία, να τους εξασφαλίσουμε αυτή την ελευθερία κυκλοφορία. Στην αρχή τους είπαμε ότι θα γίνει πριν από τα από το καλοκαίρι. Δηλαδή πληρούνται τα κριτήρια. Μετά τους είπαμε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ε, ήδη πέρασαν. Συμφωνώ κυρία Φαγιόν ότι θα πρέπει να κάνουμε έκκληση έτσι ώστε να ληφθεί αυτή η ε, απόφαση τάχιστα. Έρνεστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το προωθήσουμε όχι μόνο για λόγους νομικούς αλλά και για λόγους αρχής. Τώρα, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται όλα τα κριτήρια για τις χώρες αυτές και την εξέλιξή τους, είναι υψής της σημασία να αρθεί ε, η υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίων και να μπορέσουν να ανοίξουν προς την Ευρώπη. Και ομολογώ ότι για μένα αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από κάθε τεχνικό επιχείρημα το οποίο κατανοώ ότι είναι σημαντικό, αλλά όχι αρκετό. Βεβαίως υποστηρίζω θερμότατα την κυρία Φαγιόν. Έχει ασχοληθεί πολύ εντατικά με το θέμα. Ένα δεύτερο, το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ και με ενδιαφέρει. Αν κοιτάξουμε τώρα τα Δυτικά Βαλκάνια, έχουμε ένα μαύρο μελανό σημείο και είναι το Κόσοβο. Δεν μπορούμε να κάνουμε στην άκρη τι ζητήσει με το κοσυφοπαίδιο. Υπάρχει απόφαση του διεθνού Δικαστηρίου για το καθεστώς της χώρας και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να περιχαρακώσουμε, να περιφράξουμε τη χώρα αυτή και να μην ασχολούμαστε μαζί της. Ε, θα πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα γιατί πολύ γρήγορα θα το βρούμε μπροστά μα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα αιτήματα, δηλαδή θέλετε το λόγο. Θα ήθελα να είστε ιδιαίτερα σύντομος έτσι ώστε να ε, ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη απόψε. Ο κύριος Βαντερστούπ. Ε, ehm, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, το ε, Ολλανδικό Κόμμα της Ελευθερίας δεν χαίρεται καθόλου με την ενδεχομένη άρση θεώρησης διαβατήριων για την Αλβανία και τη Βοσνία. Και ούτε από το τελικό αποτέλεσμα είμαστε ικανοποιημένοι, ούτε από τη διαδικασία. Λέτε ότι είναι θετική τάση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι στη διεθνή διαφάνεια ε, είναι στις θέσεις 95 και 99 οι δύο χώρες, κάπου ε, τύπου Λεσότο και Ρουάντα, που είναι και πιο ψηλά ακόμα από τις δύο χώρες. Θετικές τάσεις, εντάξει, σημαίνει ότι ήταν τεράστιοι απαταιώνες και τώρα είναι μικροαπαταιώνες, αλλά απαταιώνες παραμένουν οι άνθρωποι, έτσι, αυτά μόνο. Είπα, σύντομος θα είμαι. Mr. Bronze, I'm uh, Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ χάρηκα μαθαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις Αλβανίας και Βοσνίας Ερζεγοβίνης καταπολεμούν επιτυχώς το οργανωμένο έγκλημα. Άρα αυτή η κατηγορία ανθρώπων θα μπορέσει να συνεχίσει με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες αλλού. Δηλαδή, τη στιγμή που δεν θα χρειάζονται θεωρήσεις, θα μπορούν να μεταβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 90 μέρες και ίσως και πολύ περισσότερο και να αρχίσουν την επιχείρησή τους εδώ. Άρα θα είναι πολύ καλό για το εμπόριο του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά όχι τόσο καλό για μας. Ο κύριος Κοτσέτα ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα να είσαστε ιδιαίτερα σύντομο. Εντάχει, πιστεύω ότι ότι πρέπει να πω ότι θα υπερψηφίσω την άρση της θεώρησης, αλλά θα ήθελα να πω και το εξής. Μιλάμε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και μιλάμε για την άρση της ε, θεώρησης, του καθεστώτος θεωρήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε ε, υπόψη το γεγονό ότι εκεί όπου υπάρχει ένας μαύρος κατάλογος στις χώρες αυτές, να διαβιβάζεται αυτός ο κατάλογος και προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μετακινούνται ελεύθερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει δηλαδή αυτό να αναφερθεί ρητός. Θα πρέπει να προβούμε σε μια στοχοθετημένη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος που προέρχεται από αυτές τις χώρες. Η Επιτροπή δεν χρειάζεται να απαντήσει, αλλά εάν η κυρία Μπούς το επιθυμεί, θα ακούσουμε τη γνώμη της Επιτροπής για ένα ακόμα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, με βάση τα σχόλια που ακούστηκαν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τη στιγμή που πληρούνται οι όρια για άρση της θεώρησης, τότε εμείς θα παρακολουθήσουμε την πρόοδο που επιτελείται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που επιτελείται άπαξ, αλλά ακολουθούμε τη διαδικασία διαχρονικά. Βλέπουμε δηλαδή ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν αυτές οι χώρες. Άρα η διαδικασία αυτή δεν λύγει με την έγκριση της πρότασης. Θα υπάρχει διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση προς το παρόν. Λοιπόν, και περνάμε στο επόμενο θέμα και τελευταίο που ε, συμπεριλήφθη η διάταξη μετά την απόφαση των συντονιστών που έγινε προηγουμένως. Ε, αποφασίσαμε λοιπόν να συμπεριληφθεί και αυτό το θέμα για την κατάσταση των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την κοινότητα των Ρωμά λοιπόν. Λοιπόν, θα, θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέση της στην Επιτροπή μας ε, για τη θέση της ε, ως προς τα πρόσφατα γεγονότα τον Αύγουστο. Για την κατάσταση των Ρωμά θα ακούσουμε την κυρία Φρανσουάζ Λεμπάιε, Γενική Διευθύντρια ε, της ε, διεύθυνσης, Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης που θα μας παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Λεβάη έχει το λόγο. Καλωσορίσατε ενώπιόν μας. Έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τη νέα Γενική Διευθύντρια Δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα εκφράσει εξ ονόματο. Μάλλον θέλουμε να εκφράσουμε εξ ονόματο τη Επιτροπή μα ε, όλε μα τι ευχέ για κάθε επιτυχία και ε, καλό πνεύμα συνεργασία για το έργο που έχουμε μπροστά μα. Έχετε καλό το λόγο, κύριε μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια υποδοχής και χαίρομαι για την ευκαιρία που θα έχω και προσβλέπω στη συνεργασία με την Επιτροπή σας, το πνεύμα συνεργασίας που ανέκαθεν πριτάνευε στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Ε, μου ζητήσατε να έρθω σήμερα να σας μιλήσω για τα γεγονότα και τις εξελίξεις ως προς την κατάσταση των ΡΟΜ. Μου δίνει τώρα την ευκαιρία αυτό να ενημερώσω την Επιτροπή σας για τις εξελίξεις και ε, το πώς ε, δρά και σκέπτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την ευκαιρία να εκφραστεί διαστόματος ε, της Αντιπροέδρου κυρίας Ρέντινγκ που είναι επιφορτισμένη και αρμόδια για αυτά τα θέματα. Στις 25 Αυγούστου ε, δήλωσε ότι βεβαίως τα κράτη-μέλη μπορεί ε, να ευθύνονται ε, και να φροντίζουν για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των πολιτών τους εντός της επικρατείας τους. Όταν το πράττουν αυτό όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το κάνουν σεβόμενα το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, όπως αυτά ε, περιγράφονται στο χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που θυμίζω ότι τώρα έχει και δεσμευτικό χαρακτήρα από την έγκριση και θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε την κατάσταση έτσι, από πλευράς νομικής πρώτα απ' όλα, αλλά και ε, ενσωμάτωσης και ένταξη των Ρωμά στην Ευρώπη. Για τη νομική ανάλυση υπάρχουν διάφορα στοιχεία που πρέπει να εγκρίνουμε. Βεβαίως κατά πόσο ε, τα γαλλικά μέτρα αυτά ε, συνάδουν με την οδηγία του 2004 με παριθμό 38 για την ελεύθερη κυκλοφορία είναι σαφές ότι ε, η οδηγία αυτή καθιερώνει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αλλά ε, συνοδεύεται αυτή από κάποιες προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις αυτές ποικίλουν ανάλογα με το εξής Ανάλογα αν ένας πολίτης ανούσης διαμένει σε άλλο κράτος μέλος ε, για τρεις μήνες ή πέραν των τριών μηνών. Ε, και εκεί επίσης αυτά συνοδεύονται από διάφορα διαδικαστικά μέτρα που είναι σημαντικό να σέβεται κανείς για να συμμορφούνται με την οδηγία. Και άλλο θεμελιώδες δικαίωμα είναι ακριβώς ο σεβασμός του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων αρχή της μη διάκρισης βεβαίως που είναι εγγεγραμμένη στο άρθρο 21 και είναι σημαντικό να φροντίσουμε να ελέγξουμε αν έχει γίνει σεβαστό αυτό. Γι' αυτό η Αντιπρόεδρος Ρέντιν και η κυρία Μάλστρομ ε, συνεδρίασαν με τους ε, Γάλλους Υπουργούς ε, Μετανάστευσης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για να ε, λάβουν ε, διευκρινήσεις σχετικά με το είδος των μέτρων που ελήφθησαν. Ήταν χρήσιμες αυτές οι διευκρινήσεις και πήγαιναν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάστηκε και χρειάζεται να έχουμε και περαιτέρω ε, εξηγήσει και διευκρινήσεις και γι' αυτό θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων αύριο μια συνεδρίαση με εκπροσώπους των γαλλικών αρχών. Υπό το φως όλων αυτών λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να αποφανθεί για τις νομικές πτυχές που συνδέονται με αυτό το θέμα. Ε, Παράλληλα με αυτά τα νομικά ε, θέματα είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με την κατάσταση των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ε, η Επιτροπή αυτή ασχολήθηκε με πάρα πολύ ε, μεγάλη ε, προσοχή και φροντίδα και τον Απρίλιο ενέκρινε την πρώτη δήλωση που είναι η ειδική δήλωση, η ανακοίνωση της Επιτροπής που αναφέρεται ειδικά στους Ρωμά. Παραμονές, θα θυμάστε, της Συνόδου Κορυφής της Κόρδοβα για τους Ρωμά. Και μάλιστα ε, υιοθετούσε το αντίστοιχο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είχε εγκριθεί προηγουμένως. Η ανακοίνωση αυτή συνοδευόταν και από κάποιους στόχους φιλόδοξους για ε, να ευνοηθεί η ένταξη των ε, Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι η μεγαλύτερη εθνότητα ε, στην Ένωση, 10 με 12 εκατομμύρια Ρωμά ε, ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα διάφορα κράτη-μέλη και είναι η κοινότητα εκείνη η οποία υφίσταται τις περισσότερες διακρίσεις. Γι' αυτό το λόγο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την ανακοίνωση, αλλά όχι μόνο, για το λόγο αυτό επίσης τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα διορθωτικά ταμεία, το σύνολό τους και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισφέρουν με σημαντικό τρόπο ε, για την ένταξη των Ρωμά και μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007 2013 10 δισεκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, απευθύνονται στους Ρωμά σε χώρες ιδιαίτερα που έχουν σημαντική κοινότητα αριθμητικά στην επικράτειά τους. Βεβαίως θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα αυτά που πραγματικά απευθύνονται προς τους Ρωμά ε, πραγματικά επενδύθηκαν προς όφελος εκείνων ε, των ε, προσώπων της κοινότητας των Ρωμά. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της προέβλεψε συνόδους κορυφής υψηλού επίπεδου δηλαδή με τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως. Έχει γίνει μια τέτοια συνάντηση με την Ουγγαρία νωρίτερα φέτος και μια δεύτερη σύνοδος κορυφής θα ακολουθήσει τον Οκτώβριο με τη Ρουμανία. Στόχος είναι να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη που θα το χρειαστούν για να βεβαιωθούμε ότι ε, θα υλοποιηθούν και θα εκτελεστούν τα σωστά έργα για την κοινότητα αυτή, γιατί είναι περίπλοκα τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα αυτή. Ε, είναι προβλήματα παιδείας, προβλήματα που συνδέονται με την υγεία, με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό χρειάζεται συντονισμένη δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, εκτελεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, έμπνευση του Κοινοβουλίου κατά για να ενταχθεί η κοινότητα αυτή και, και να ακολουθεί μία μέθοδος συγκεκριμένη για να μπορούν να ενταχθούν οι Ρωμά στις κοινωνίες μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκε βεβαίως υπό το πνεύμα αυτό με τις ρουμανικές αρχές για να συζητήσει και ε, να δει ποιες είναι οι προθέσεις της Ρουμανίας ως προς την ένταξη, την ενσωμάτωση των Ρωμα και να βεβαιωθεί ότι διατηρείται η προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχουν δυσκολίες ένταξης του Ρωμά ε, στην κοινωνία και δήλωσε προθυμία να ε, συμμετέχει ως ειλικρινής και ήμιος διαμεσολαβητής για να ενισχυθούν τα μέτρα στα κράτη-μέλη που απευθύνονται στην κοινότητα το Ρώμα και πιο συγκεκριμένα στην ε, συμπεριλήψή τους και στην ένταξή τους. Και με τον ίδιο επίσης τρόπο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο γιατί ακριβώς εκεί ε, ε, στις περιφέρειες ε, χρειάζονται τα μέτρα πιο κοντά στους Ρωμά. Αυτά. Έτσι έχει η κατάσταση των πραγμάτων, ο προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω συνεχίζεται η προσπάθεια και η εξέταση και των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την ευκαιρία να ακούσει την παρουσίαση της Επιτρόπου κυρίας Ρέντινγκ, της Αντιπροέδρου, μετά τις επαφές που θα έχουν μεσολαβήσει με τη γαλλική κυβέρνηση. Euh, euh, και συνεχίζει το προβληματισμός και η περισυλλογή για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινότητες των Ρωμά θα ενταχθούν στην κοινωνία. Είναι πραγματικά μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το σύνολο της Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λεμπάιλ. Ε, σας ε, θυμίζω όλους πόσο σημαντικό είναι να τηρηθούν τα χρονικά όρια. Δηλαδή 6,5, 18 και 30 είναι το τέλος της συνεδριάσεως. Άρα έχουμε λοιπόν περίπου 30 λεπτά για 20 σχεδόν παρεμβάσεις. Υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός ε, των μελών της Επιτροπής που έχουν ζητήσει τον λόγο. Παρακαλώ λοιπόν να συμβάλλετε όλοι στο να τηρηθούν τα όρια του χρόνου. Ε, εγώ θα σας σημάνω το τέλος ε, του χρόνου ε, παρεμβάσεώς σας που θα είναι ενός λεπτού. Κύριε Μπουσούτιλ, πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση. πότε θα είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει άποψη σχετικά με το εάν η Γαλλία συμμορφώνεται με το ε, κοινοτικό δίκαιο σχετικά με τα όσα τεκταίνονται στην χώρα αυτή. Ε, θα γίνει η συζήτηση την επόμενη εβδομάδα, στην περίοδο συνόδου. Θα ήταν καλό να έχουμε τη δήλωση αυτή πριν από την ε, συζήτηση αυτή. Κύριε Μωράς. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομος. Στην δήλωσή σας κυρία Διευθύντρια μιλήσατε για την εφαρμογή της ανακοινώσεως της Επιτροπής της, ε, του Απριλίου και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνικοπολιτική θέση των ε, ΡΟΜ. Αυτό που θα χρειαστεί να απαντηθεί για την επόμενη εβδομάδα είναι πρώτο η προσωρινή έκθεση θα καλύψει τα όσα πρόκειται να πω. Θα έχει κάποια πολιτική επίδραση, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, όρια για την ελευθερία διακίνηση ε, των Ευρωπαίων πολιτών και η οδηγία τα προβλέπει αυτά. Θα φτάσει μέχρι το θεμελιώδες θέμα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται για ολόκληρη ομάδα προσώπων που ενδεχομένως ε, απελάβνεται συλλογικά και επομένως δεν υπάρχει περιθώριο για την ατομική αντιμετώπιση των ατομικών αυτών περιπτώσεων που ε, προβλέπεται στο νόμο. Η κυρία Ρέντιν και οι άλλοι δύο επίτροποι είναι διατεθειμένοι να ε, θέσουν ακριβώς αυτό το θέμα. Η κυρία Εντφέλτ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ το θέμα, γιατί συχνά έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ διστακτική. Νομίζω όμως τώρα είστε, βρίσκεστε στον έλεγχο της καταστάσεως και θα παρέμβετε εάν χρειαστεί. Αυτή την εντύπωση έχω. Όπως ο κύριος Μπουσουτήλ θα ήθελα να μάθω και εγώ αν θα μπορέσετε να μας ενημερώσετε πριν να διεξαγάγουμε τη συζήτησή μας. Θέλω να μάθω επίσης όμως εάν προτίθεστε να δεχθείτε την πρόσκληση της γαλλικής κυβερνήσεως για συμμετοχή σε συνεδρία στην επόμενη Δευτέρα νομίζω, διότι οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να οργανώσει όποια συνεδρίαση θέλει και να προσκαλέσει όποιον θέλει. Αλλά πιστεύω ακόμη ότι είναι λίγο παράξενο ότι αυτό συμβαίνει εκτός πλαισίου Ευρωπαϊκής ενώσεως. Ενώ υπάρχουν εν προκειμένου θέματα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι θα ήταν λάθος το μήνυμα εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέλθει σε τέτοια συνεδρίαση. Η κυρία Φλότχε. Σας ευχαριστώ. Και εμένα με ικανοποιεί η παρουσία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και η επαγρυπνησή της. Θεωρώ ότι ο ρόλος της είναι του θεματοφύλακος των συνθήκων και ότι η υπόθεση αυτή άπτεται των θεμελιωδών και συνταγματικών ελευθεριών ε, που προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, της ελευθερίας διακίνησης και της ισότητας των Ευρωπαίων πολιτών ενώπιον του δικαίου. Από την άποψη αυτή νομίζω ότι ασφαλώς πρέπει να υπερβείτε τα όρια μιας, ενός ακροβατικού εγχειρήματο που κάνει η γαλλική κυβέρνηση και που ήδη αμφισβητούνται και ενώπιον της ε, γαλλικής, και γαλλικής δικαιοσύνης και να εξετάσετε πιο κοντά, από πιο κοντά αυτή την έννοια της ε, ε παραβίασης της δημόσιας τάξης που προκάλεσε και δήλωση της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η θλιβερή υπόθεση θα οδηγήσει σε μια μεγάλη κίνηση για ένταξη, για ενσωμάτωση των ε, ΡΟΜ στην, ευρωπαϊκή, στην κοινωνία, στη ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλο δυναμισμό, με μεγάλη ε, θεληματικότητα όπου θα πρέπει να δείξει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι η θεματοφύλαξη των ευρωπαϊκών συνθήκων όποιοι και όποιες και είναι οι λαϊκιστικές απόψεις στις διάφορες χώρες. Ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι που ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εργάζεται τόσο εντατικά για το θέμα. Αλλά ολόκληρο το καλοκαίρι, παρατηρώντας ε, προσεκτικά από τον τύπο τι συνέβαινε στην Γαλλία, είχαμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν διστακτική. Και όταν έγιναν κάποιες πρώτες δηλώσεις, ε, μίλησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για και για εθνικές αρμοδιότητες. Ενώ πρόκειται για θεμελιώδη θέματα, δηλαδή θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι απόλυτα παραδεκτά αυτά. Έχω και μια ερώτηση. Το κοινοβούλιο ζήτησε κατ' επανάληψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να καταθέσει μια ε, συνολική ευρωπαϊκή στατική για την ένταξη των ΡΟΜ. Τώρα το θέμα αυτό λαμβάνει ακόμα πιο επίγοντα και σημαντικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς το βλέπετε το πράγμα αυτό και πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τέτοιου είδους στρατηγική. Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι που συζητούμε το θέμα αυτό ή τουλάχιστον το θίγουμε. Θα είμαι σύντομη, αν και είμαι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη με τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Όχι όμως μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες. Αυτό εν παρενθέσει. Τώρα, έχω νομικά ερωτήματα. Δεν είναι καταρχήν παραβίαση του δικαίου όταν γίνονται συλλογικές απελάσεις χωρίς εξέταση της μεμονωμένης περίπτωσης. Δεύτερο, δεν ε, παραβιάζεται η αρχή απαγόρευσης των διακρίσεων με αυτή την ε, αντιμετώπιση. Τέλος, η οδηγία περί ελεύθερης διακίνησης. Επίσης θεωρώ ότι παραβιάζεται. Και επίσης μ, ε, ρωτώ πότε θα υπάρξει, όπως και η κυρία Γκρινγκό, αυτή η περίφημη στρατηγική για την ένταξη των ΡΟΜ. Ελπίζω ότι με την αφορμή αυτή θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξής. θα αποφανθεί για αυτή την παραβίαση των δικαιωμάτων του χάρτη. Γιατί είναι παράδοξο να μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένταξη. Ποια ένταξη, αφού τους απελάβνουν. Έλαση μιας μειονότητας. Και ζητάνε από κάποιους άλλους να τους εντάξουν στις κοινωνίες τους. Μα ποιες χώρες θα εντάξουν κάποιους ανθρώπους που κάποια ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελάβνουν. Παράδοξο δεν είναι, για να μην πω υποκριτικό σχεδόν. Νεκρό γράμμα έχει καταντήσει ή έχουμε καταντήσει το χάρτη. Δεν είναι ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό θα ήταν αν εξεταζόταν περίπτωση κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Και ξέρετε δεν το κάνει μόνο η κυβέρνηση Σαρκοζή και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρχίζουν αυτές τις διαδικασίες. Και έχουμε ένα μέγα δράμα, ένα κύμα ρατσισμού που διαπερνά την Ευρώπη ολόκληρη. Και αν δεν λάβει τώρα μέτρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποια στιγμή μπορεί να είναι πολύ αργά. Αυτή λοιπόν την ερώτηση ήθελα να σας υποβάλω. Τι θέση θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριος Μίλντορ. Σύντομος και εγώ ευχαριστώ για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το μείζον νομικό πρόβλημα εδώ. Είναι ο συλλογικό χαρακτήρας των δράσεων αυτών. Τα ίδια τα γαλλικά δικαστήρια τώρα εξετάζουν το θέμα. Δεύτερο υπό την παρούσα δημοσιονομική προοπτική πρόκειται να δαπανηθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε βρεθεί, βρισκόμαστε τώρα στα μισά περίπου. Ποιε είναι οι πρώτε δράσει που έχουν αναλυθεί με αυτά τα χρήματα. Ένσιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι ενέργειες της γαλλικής κυβερνήσεως είναι στην ουσία απέλαση και δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε. Θα ήθελα να πω ότι η εθνο, εθνότητα των Ρώμα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να γίνουν κατανοητές. Και μόνο όταν τις κατανοήσουμε τότε μόνο θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ένταξή τους. Το λάθος που έγινε είναι ότι οι Ρώμ δεν θεωρήθηκαν Ευρωπαίοι πολίτες με τα αρμόζοντα δικαιώματα, αλλά ως μετανάστες και τους φέρθηκαν με τον τρόπο αυτό ενώ η αντιμετώπιση τους θα πρέπει να αποτελέσει, ε, ε, θα πρέπει να ενταχθεί μάλλον σε μια στρατηγική συνολικότερη ένταξή του. Η υπόθεση των ΡΟΜ πρέπει να επανεξεταστεί στα πλαίσια μιας επίγουσας μελέτης. Θα μου πείτε ότι έχουν γίνει πολλές ήδη μελέτες, αλλά οι μελέτες αυτές ή ήταν ατελείς ή τα πορίσματά τους ήταν εσφαλμένα. Βεβαίως και οι έχουν, οι Ρομ έχουν ανάγκη ε, να ενσωματωθούν, αλλά όχι με τη βία. Σας ευχαριστώ. Τάις. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μας κάνει εντύπωση ε, στη συζήτηση η ε, υπερβολικές αντιδράσεις των συναδέλφων. Μιλάνε για απέλαση, για ρατσισμό, αμέσως εξάπτονται. Μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε σχέση και με το κοινό αίσθημα των πολιτών, να μην χάσουμε την επαφή μας. Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Ε, πήρε μέτρα η Γαλλία γιατί υπάρχουν προβλήματα και κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι, ευρωπαϊκοί κανόνες νομίζω που να έχουν παριαστεί. Ήταν αναπερίπτωση ε, εξέταση κάθε φακέλου, κάθε προσώπου υπήρχαν παράνομοι άνθρωποι που είχαν παράνομους καταβλισμούς ε, μεγάλα προβλήματα προκλήθηκαν, ε, διαπιστώθηκε εγκληματικότητα, παραβατικότητα και αντέδρασε η γαλλική κυβέρνηση και έχει το δικαίωμα εντό τη επικουρικότητα και τη εθνική κυριαρχία κάθε κράτου μέλου. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο γίνεται λιγότερο, να κατεβόμαστε εκεί μέσα. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμε. Indeed, we are facing a problem which is a European problem. Πράγματι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Με ευρωπαίους πολίτες, τους ΡΟΜ, με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ευρωπαϊκό δίκαιο και ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες. Η κυβέρνηση του Πρόεδρου Σαρκοζή υπερεύει τα εσκαμμένα κατά τρόπο προκαλεί αγανάκτηση δίνοντας έτσι αφορμή στην ανάπτυξη ξενοφοβίας και ρατσισμού Πρόκειται για συλλογική απέλαση και συλλογικό στίγμα εγκληματικότητας. Βλέπουμε τον Υπουργό Ορτεφέ να μιλεί για στατιστικές εγκληματικότητας που ε, είναι λέει χαρακτηριστικό των Ρουμάνων, όχι των Ρωμ. Να λοιπόν οι συγχύσεις πώς προκύπτουν δεν μιλούμε εδώ για ενσωμάτωση. Έχουμε καλό παράδειγμα ενσωμάτωση στον ΡΟΜ που είναι η Ισπανία. Η ενσωμάτωση όμως δεν μπορεί να γίνει εάν για παράδειγμα αντιδρούν οι αρχές των χωρών υποδοχής. Θα ρωτήσω λοιπόν την Κομισιόν τι μπορεί να μας πει σχετικά με την αντίδραση του Πρόεδρου Μπασέσκου στη Ρουμανία που έκανε πολύ ε, δυσάρεστα σχόλια σχετικά με τον πληθυσμό των ΡΟΜ. Η Κομισιόν, εκτός από έντιμος διαμεσολαβητής, είναι και θεματοφύλακα των συνθήκων. Και ρωτώ λοιπόν, είναι διατεθειμένη η Κομισιόν να αναλάβει δράση για να καταγγείλει και την κυβέρνηση του πρόεδρου Σαρκοζή και, τον, και τις άλλες κυβερνήσεις που έδρασαν με τρόπο απαράδεκτο όπου όπως είπε ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας Μαδούρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αποτελεί παραβίαση της συνθήκης της Λισαβόνας. Η κυρία Βεργία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γενική Διευθύντρια, επιτρέψτε μου να δώσω μερικά αριθμητικά στοιχεία για τη γαλλική πραγματικότητα, για να μπορέσει ο καθένας να δει στο σωστό πλαίσιο το θέμα, να το σχετικοποιήσει. 36.000 Ρωμά ζουν στη Γαλλία, 850.000 στην Ισπανία και 650.000 στην Ιταλία, ε, βουλγαρικής και ρουμανικής καταγωγής. Γι' αυτό τα λόγια του Προέδρου Σαρκοζή είναι ιδιαίτερως απαράδεκτα. Θα πρέπει να πούμε ότι η γαλλική κυβέρνηση ε, θέλει να ε, δείξει ε, ότι κάνει απελάσεις μαζικά 25 με 30 χιλιάδες το χρόνο και θέλει να έχει αποτέλεσμα ποσοτικό για να καταπολεμήσει τη λαθρομετανάστευση και ε, από αυτούς είναι ε, οι 6 έως 9 χιλιάδες Ρουμάνοι το 1 τέταρτο των απελάσεων των υποτιθέμενων αλλοδαπών εντός εισαγωγικών στη Γαλλία είναι Ευρωπαίοι πολίτες Ρωμά και είναι πρακτικό να του διώχνεις γιατί ξανάρχονται κάθε τρει μήνε και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λογιστικού σκοπού πολλέ φορέ το χρόνο. Και αυτό εξηγεί ε, και ε, τη στάση της κυβέρνησης και την αντίσταση απέναντι στη ρουμανική κυβέρνηση. Οι καταβλισμοί τους ε, διώκονται από την αστυνομία με τρόπο συνοπτικό στις διαδικασίες. Πώς να γίνει ανάλυση σε ένα περίπτωση. Ε, έρχονται με έτοιμα τα έγγραφα οι αστυνόμοι. Με ε, κλήσεις και παραβάσεις και προφανώς είναι μαζικές απελάσεις. Και θα ήθελα να ε, απευθυνθώ στον κύριο Μπουσουτήλ και να πω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ησυχία της ήρεμα να εξετάσει τη γαλλική πραγματικότητα και να ακούσει τις οργανώσεις των πολιτών ε, που συνεργάζονται με τους Ρωμό και κάνουν ε, καταπληκτική δουλειά και με αριθμητικά στοιχεία έχουν ε, εκδώσει μια έκθεση, την έχουν στείλει σε όλους τους βουλευτές και ελπίζω να την έχουν απευθύνει και εσά. Ευχαριστώ. κυρία Μπορσελίνο. Grazie, grazie alla direttrice generale. Ευχαριστώ την ε, Γενική Διευθύντρια. Βεβαίως είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Οι συνθήκες παραβιάστηκαν και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευρωπαίοι πολίτες που υφίστανται διακρίσεις με βάση την ε, εθνική τους ε, προέλευση, όχι με βάση τη συμπεριφορά τους ή την εδώ θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή λοιπόν στα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία και αυτά που πράττει η κυβέρνηση Σαρκοζή. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Ιταλία, όχι με την ίδια έκταση, αλλά και με προληπτικό τρόπο ε, στην Ιταλία. Και οι Ρουμάνοι πολίτες διώχθηκαν πάλι ε, με ε, επιθέσεις κατά καταβλισμών Ρωμά και με ρατσιστικό μίσος και μένος που βρήκε πολύ έντονη έκφραση στην Ιταλία και βεβαίως ο τύπος δεν παρέλειψε να ε, δώσει ε, μεγάλη προβολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέτε ενδιαφέρθηκε. Ναι, μπορεί να ενδιαφέρθηκε τώρα, αλλά στην αρχή ήταν πάρα πολύ ε, δειλή η αντίδρασή της. Τώρα επήγει η αντίδραση και χρειάζεται ε, πραγματικά να ληφθούν μέτρα για την ένταξη, την εσωμάτωσή του. Άρα δεν ήταν ενταγμένοι στην κοινωνία. Και πού πήγαν τα κονδύλια αυτά. Υπάρχει κίνδυνος τώρα ε, να επεκταθεί η κατάσταση και σε άλλες χώρες. Και ο κύριο Μαρόνι κάνει ήδη δηλώσει στην Ιταλία. Ευχαριστώ κύριε Κέλλε. Στην περίπτωση όπου διαπιστώσετε ότι οι απελάσεις αυτές παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο και εγώ είμαι βεβαία γι' αυτό. Τι ακριβώς, ε, πώς ακριβώς μπορείτε να αντιδράσετε στις ενέργειες της γαλλικής κυβερνήσεως και των άλλων κυβερνήσεων. Μάλιστα, ευχαριστώ. Η κυρία Πράγματι, η ΡΟΜ στη Γαλλία είναι ένας χρήσιμος αποδιοπομπαίο τράγος για την παρούσα κυβέρνηση Δύο ερωτήσεις τώρα. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συνέχεια σκοπεύει να δώσει κυρίως στο κείμενο του προηγουμένου Μαρτίου του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να μπούμε σε ένα νέο στάδιο που θα είναι λιγότερο αμυντικό αλλά και πιο συντονισμένο για να αντιμετωπιστούν με ευνοϊκότερο τρόπο η ΡΟΜ. Δεύτερο, ποιες είναι οι προθέσεις της Κομισιόν για να διασφαλίσει ώστε οι διάφορες ενδιαφερόμενες χώρες, δεν είναι μόνο η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Γαλλία, εδώ και τελευταίες εβδομάδες ε, βρίσκονται στην επικαιρότητα, να τεθούν ενώπιον των ευθυνών του και απέναντι στο ευρωπαϊκό δίκαιο και απέναντι βέβαια στην ανάγκη ένταξη συμπερίληψη των ε, ΡΟΜ. Ο κύριος Βάντερ Στούπ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον παρακαθήμανο ότι είναι γελία αυτά τα μεγαλόστομα που ακούμε εδώ. Το, το κοινοβούλιο έχει εξαγριωθεί και ε, στρέφεται κατά ενός κράτους που επιβάλλει τον νόμο. Και εγώ δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση ε, στη Γαλλία, αλλά στην Ολλανδία ξέρω πολύ καλά ότι τα τρία τέταρτα το Ρωμά έχει ποινικό μητρό. Και ο Υπουργός Φαντελάν, σοσιαλιστής, είπε ότι ε, ε, οι ίδιοι οι Ρωμά θέτουν σε αυτούς τους εκτός της κοινωνίας. Σοσιαλιστής υπουργό το είπε αυτό. Μα εμείς δεν έχουμε δουλειά τώρα να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Είμαστε εκτός θέματος. Είναι θέμα της Γαλλίας. Εγώ θεωρώ ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να απελάβνεται και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν συμφωνώ με την αριστερή πλευρά του σώματος. Ε, να διευρυνθεί η δυνατότητα αυτή, όχι να περιοριστεί. Λοιπόν, αφήστε τη Γαλλία να κάνει αυτό που πρέπει και εμεί να μην ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. 20 μέλη έλαβαν το λόγο σε 25 λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής μας να μας δώσετε πάνω, ε, ε, ε, το πολύ πέντε λεπτά για να μας απαντήσει η κυρία Λεμπάρ, Γενική Διευθύντρια ε, Δικαιοσύνης Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέντε λεπτά για να απαντήσω σε 20 ε, παρεμβάσεις δεν είναι πολλά. Ε, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ομαδοποιήσω ε, τις παρεμβάσεις. Ε, φαίνεται η πολυπλοκότητα του προβλήματος από τόσα είπατε. Δεν είναι καθόλου απλό και θα πρέπει να ειδωθεί από πολλές πτυχές και οπτικές γωνίες. Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων έχει να κάνει με τη νομική κατάσταση. Αυτό που μπορώ να σας επαναλάβω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θέματοφύλακας των συνδικών και υπεύθυνη ε, να εφαρμόζεται σωστά από τα κράτη-μέλη το κοινοτικό δίκαιο οι συνεδριάσεις που έγιναν με τις γαλλικές αρχές έχουν ως στόχο ακριβώς να διαπιστώσουν τα πραγματικά περιστατικά και να αποκομίσουν διευκρινήσεις, δηλαδή να γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση και από τη σκοπιά της ελεύθερης διακίνησης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και Τη μη διάκριση να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, τι συμβαίνει. Αυτό πρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχιστεί και αύριο σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων και τεχνικό επίπεδο με τι γαλλικέ αρχέ. Ε, άλλη ερώτηση που κάνατε πολύ, πότε θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μόλις έχει πλήρη γνώση της κατάστασης θα αποφανθεί. Η αυριανή λοιπόν συνεδρίαση θα είναι χρήσιμη και την άλλη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακούσει την κυρία Ρέντινγκ, την Αντιπρόεδρο ε, που θα παρουσιάσει ε, την κατάσταση με τις διευκρινήσεις και τις εξηγήσεις που θελήσαμε να μας δώσουν οι γαλλικές αρχές και το συντομότερο θα αποφανθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η συζήτηση της επόμενης εβδομάδας σίγουρα αποτελεί ευκαιρία να γίνει κάτι τέτοιο. Μια άλλη ομάδα ερωτήσεων έχει να κάνει με τα κονδύλια και τις πιστώσεις για την ένταξη των Ρωμά, 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι απέγιναν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι είναι στη ε, διαχείριση τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι βασική ευθύνη των κρατών μελών δηλαδή να εκτελούν τα προγράμματα και τα έργα, αλλά βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρακολουθεί αυτά τα θέματα και το συζητήσαμε συνεδριάσεις με ε, τους Ρουμάνους. Να δούμε πώς υλοποιούνται τα προγράμματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υποστηρίξει τα κράτη-μέλη που το ζήτησαν για να τα βοηθήσει να ε, βρουν ποια θα ήταν εκείνα τα έργα που θα χρησιμεύαν προς την κατεύθυνση αυτή. Και είναι βεβαίως πρόθυμη και διατεθειμένη να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε επίση μια ερώτηση για την ιδιαιτερότητα το όνομα για τον διάζοντα χαρακτήρα και βέβαια λαμβάνονται αυτά υπόψη. Εξού και είναι περίπλοκο το θέμα για να βρούμε σωστές λύσεις, τις καλές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζεται λοιπόν ο προβληματισμός, επαναλαμβάνω, και η περισυλλογή και για τη νομική πτυχή αλλά και τα μέσα ένταξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνω, θα ακούσει την αφορά της κυρίας Ρέντιν και θα συμμετέχει και στις δικές σας συζητήσεις στην Ολομέλεια. Κάτι ακόμα ως διευκρίνηση για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την παρουσία της στην ε, συνεδρίαση που διοργανώνουν οι Γάλλοι οι γαλλικές αρχές για ε, ορισμένους υπουργούς εσωτερικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκληθεί στη συνεδρίαση αυτή και η αρμόδια επίτροπος που είναι η κυρία Μάλστρομ ε, αρμόδια για τα θέματα εσωτερικών ε, υποθέσεων θα συμμετέχει και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθύντρια και για την ενημέρωση σας προσφέρω τις καλύτερες ευχές μας για, το, για τη μελλοντική σας εργασία. Ευχαριστώ και τους Γερμηνείς και ε, καλό σας βράδυ.